Κυρίες και κύριοι, έστω βράδυ απεβίωσε ο επί συναδελφός μας, ο κύριος Βίλφρεντ Μαρτάνς, ο οποίος είχε γεννηθεί τον Απρίλιο 1936 και ήταν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Είχε μεγάλη σταδιοδρομία στο Βέλγιο, στο ευρωπαϊκό επίπεδο και εδώ πέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο κύριος Μάρτενς από το 1979 μέχρι το 1992 με μικρά διαλύματα ήταν πρωθυπουργός του Βελγίου. Από το 1994 μέχρι το 1999 ήταν επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ο Βίλφιντ Μαρτένς ήταν βαθύτατα πεπισμένος Ευρωπαίος ολόκληρη την πολιτική της ζωή την αφιέρωσε στην υπηρεσία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ήταν ένας εξαιρετικός εκπρόσωπος της κοινότητας Μπενελούξ. Η ίδρυση της οποίας ήταν κομμάτι της ίδρυσης των ευρωπαϊκών κοινοτήτων και η συνεισφορά της ε, οποίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανεκτήμητη. Ο κύριος Μάρτενς ήταν επίσης βαθύτατα καθολικός γιατί αντιλαμβάνονταν την κοινωνική διάσταση του καθολικισμού και ήταν εξαιρετικός πολιτικός του χριστιανοδημοκρατικού κινήματος στην Ευρώπη. Αλλά αυτό το οποίο πάντα έλεγε ήταν πως η συνεισφορά των εθνικών κρατών στη μεταπολεμική Ευρώπη πρέπει να είναι στο να ξεπεράσουμε τους διχασμούς σε αυτή την Ήπειρο μέσω της συνεργασίας λαών και κρατών γιατί το μήνυμα που λαμβάναν πάντα ήταν πως η Ευρώπη είναι ενωμένη όταν, ε, όταν είναι ισχυρή όταν είναι ενωμένη. Αν λοιπόν δεχτούμε το μήνυμα του Βλήφρετ Μαρτένς για το σεβασμό και για το γνώμη του άλλου θα είναι σε καλό δρόμο η Ευρώπη. Στο πρόσωπο του Βίλφρεντ Μαρτένς, οι συνάδελφοι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος χάνουν έναν εξαιρετικό ηγέτη το δε βασίλειο του Βελγίου έναν μεγάλο Βέλγο και η Ευρωπαϊκή Ένωση χάνει έναν μεγάλο Ευρωπαίο. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή προς μήν του Βίλφετ Μαρτένς. sie haben sich zu ehren von wilfried martens von ihren plätzen erhoben. ich danke ihnen. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι μεγάλη χαρά για εμένα, είναι τιμή κυρίες και κύριοι το ότι μπορώ να σας αναφέρω